Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές μας ενημέρωσαν για την εκλογή του Άρεντ Κον στη θέση του Μάρτιν Σούλτς από την 24η Φεβρουαρίου 17. Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν την εκλογή του κυρίου Κον, τον καλωσορίζουμε.